Colegi, putem trece la explicațiile de vot. Ακολουθούν επεξηγήσεις ψήφου τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Συνεχίζεται η συζήτηση. Παρακαλώ, έχουμε τις επεξηγήσεις ψήφου τώρα. Ραπόρτο Μαριέλ Δεσάρνεζ, δάω κουβέντου δόμνului Καπούτο. Λοιπόν, έκθεση Δεσάρνεζ, ο λόγο έχει ο κύριος Καπούτο.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 Ε, πληγή από την αρρώστια της ξυλέλα. Και είπαμε ότι το 2015 είχαμε εισαγωγές από την Τινησία στην Αιτία που έχουν αυξηθεί ε, 40% ή 400%. Οπότε είπαμε ότι έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες τόνων οι οποίοι θα εισρεύσουν λόγω της ε, συμφωνίας σύνθεσης και βλέπουμε ότι θα έχουμε επιπλέον άλλους 90.000 τόνους και έτσι βλέπουμε ότι θα υπάρχει φτωχοποίηση και περισσότερες απάτες. Και είπαμε ότι τώρα θα υπάρξει αθέμητος ανταγωνισμός σε σχέση με την ευρωπαϊκή ποιότητα. Είπαμε να υπάρξει ε, υποστήριξη της οικονομίας της νησίας, αλλά πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο. Δεν θα είναι δυνατόν η παραγωγή του ελαιολάδου να πληρώσουν την ύφη. Πρόεδρος, είναι το λόγο στον κύριο Γκέλνης. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο, Πρόεδρε. Έχω την εντύπωση ότι δεν βγαίνει η γαλλική διερμηνία. Δεν ξέρω, κάποιο τεχνικό πρόβλημα υπάρχει. Δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω ε, τα όσα μας εξέθεσε ο συνάδελφος μόλις. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. Ζητώ συγγνώμη, θα ελέγξουμε αυτό το τεχνικό πρόβλημα και θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε. κύριος Χάναν. σάλα. Αποσιάζει. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Από τη μια είναι μεγάλη η χαρά μας για την έκθεση που εγκρίθηκε γιατί η καλύτερη αναπτυξιακή βοήθεια είναι το αμοιβαίο εμπόριο. Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών ε, που σημαίνει οικονομική ανάπτυξη και αυτό σημαίνει θέσεις εργασία. Θέσεις εργασία σημαίνουν ε, εισόδημα και ευημερία. Μέχρι εδώ καλά. Ωστόσο γνωρίζουμε από την άλλη στι ποσοστώσει των γεωργικών προϊόντων ότι υπάρχουν παράπλευρες απώλειες ε, στην εσωτερική αγορά. Θα πρέπει να το προσέχουμε και να το λέμε και στα οποροκυπευτικά ακριβώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε υποβόσκους υπερπαραγωγή και ε, μπορεί να μειωθεί το εισόδημα ε, των παραγωγών μας όσο μικρή και αν είναι η ποσότητα ενός περιόδου που εισάγονται. Παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτον να τα έχει υπόψη της αυτά και δεύτερον να σκεφτεί αντισταθμιστικά μέτρα για τους Ευρωπαίους αγρότες. Ευχαριστώ και εμείς ευχαριστούμε λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Τάκουλα. Χάνου, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω για τη συνεργασία μας με την την Ισία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να την υποστηρίξουμε τη χώρα αυτή, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ε, τη μετάβασή της στη δημοκρατία. Στη Βόρεια Αφρική χρειάζεται να σταθεροποιηθεί η δημοκρατία και όχι μόνο στη Βόρεια, σε όλη την Ήπειρο. Δεν θα πρέπει όμως να ξεχάσουμε και τους δικούς μας ελαιοπαραγωγούς στη Νότια Ευρώπη, να διατηρηθεί η παραγωγή και να έχουμε υπόψη μας πάντα την ποιοτική παραγωγή ε, ελαιολάδου στη Νότια Ευρώπη. Τώρα που αποφασίστηκε αυτή η ποσόστοση ατασμολόγητη, ε, τι να κάνουμε. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να έχει αυξηθεί, αρκούσε η ποσότητα. Συμφωνώ με τον κύριο Καπούτο. Ευχαριστώ. Προχωράμε στην έκθεση κυρίας Γκροστέτ. Ο κύριος Μαμίκινς έχει το λόγο. Ε, ε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για μια πρόταση η οποία αποτελεί απόπειρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσει σε νομοθέτηση για τα προβλήματα της υγείας των ζώων. Οπότε θα πρέπει να δούμε ότι τώρα έχουμε νέα φάρμακα και για τα ζώα όπως και για τους ανθρώπους. Οπότε με αυτό το σχέδιο ψηφίσματος θα βελτιωθεί η πρόσβαση στα υπάρχοντα φάρμακα. Επίσης θα δοθούν κίνητρα για καινοτομία και ανάπτυξη για νέα φάρμακα. Επίσης θα καταπολεμήσουμε την ανθεκτικότητα των βακτηρίων. Εγώ ψήφισα υπέρ στην ψηφοφορία που έγινε στην Ολομέλεια. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η Γεωργία ανταποκρίνεται στις ευθύνες της. Και στα κτηνιατρικά φάρμακα πρέπει να προσέξουμε τα εξή δύο. Πρώτον, θα πρέπει να είναι λελογισμένη η χρήση και να προσανατολίζεται στην ευημερία των ζώων. Και δεύτερον, θα πρέπει να κοιτάμε τις παρενέργειες ε, για τον άνθρωπο. Βλέπε αντίσταση στα αντιβιωτικά. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε κάποια αντιβιωτικά τα οποία να είναι ένα είδος ε, εφεδρείας και να μην χρησιμοποιούνται στα ζώα παρά μόνο στον άνθρωπο. Αυτό είναι ένα τμήμα μόνο του προβλήματος και πρέπει να το γνωρίζουμε. Με την έκθεση αυτή ε, βρίσκουμε καλούς συμβιβασμούς Θέλουμε να απαγορεύσουμε το ιντερνετικό εμπόριο αντιβιωτικών και να περιορίσουμε στο ελάχιστο τη χρήση ε, και να υπάρχει διαδικασία διπλής έγκρισης η οποία υιοθετείται για τα ε, εφεδρικά ε, αντιβιωτικά γιατί είναι πολύ σημαντικό να περιορίζεται η χρήση τους και να χρησιμοποιούνται μόνο στον άνθρωπο. Ευχαριστώ. Προχωρούμε τώρα στην έκθεση Τανασέσκου. Ο κύριος Πόσπης έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Αυτό συνδέεται με το προηγούμενο ε, σημείο και σχετίζεται με τα κτηνιατρικά φάρμακα. Χαίρομαι που ε, μία οδηγία πλέον ε, είναι ο τρόπος που διαλέξαμε για να ρυθμίσουμε αυτά τα ζητήματα. Νομίζω ότι είναι σωστή η προσέγγιση. Έτσι στο μέλλον μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα έχουμε καλύτερα κτηνιατρικά φάρμακα. Νομίζω ότι αυτή, αυτό είναι το βασικό πνεύμα της έκθεσης ε, και γι' αυτό θα την υποστηρίξω. Παρατηρώ με ικανοποίηση ότι υιοθετούμε θετική προσέγγιση για, αυτή την, για αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Πρόεδρος. Παρακαλώ. Καλωσορίζω της, ε, τη νέα προσέγγιση για την χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Ε, θεωρώ επίσης ότι ο ρόλος ε, της υπηρεσίας για την καταγραφή στα μητρώα των ιατρικών φαρμάκων είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση τώρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε χωριστά εθνικά συστήματα, χρειαζόμαστε ένα κοινό παρονομαστή, καλωσορίζω. Οποιασδήποτε αλλαγέ περιορίζουν την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θέλω να λειτουργούμε βάσει βάση εκτελεστικών πράξεων, αλλά με συναπόφαση. Είναι πολύ καλό επίσης που θα γίνεται αναθεώρηση κάθε πέντε χρόνια. Αυτό και υπερψήφισα. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμπληρωματικά προς την προηγούμενη έκθεση ε, θέλω να πω το εξή. Καταρχήν δεν μπορεί κανείς να συμφωνήσει με την παρούσα έκθεση. Θέλω να πω ότι χαίρομαι που η γεωργία είναι τόσο διαφανής εδώ και με τέτοια ε, ε πυκνότητα απόδειξης και με τις νέες ε, διαδικασίες αδειοδότησης και έγκρισης για τα κτηνιατρικά και θα παρακαλούσα όλα αυτά που έχουμε επιβάλει στη Γεωργία και αυτή την κατάσταση να τη μεταφέρουμε και στην ανθρώπινη ιατρική. Διότι δυστυχώς σήμερα σε ό,τι αφορά την ενημέρωση ε, της μεθόδους θεραπείας και τη χορήγηση πολλά είναι σε γκρίζες ζώνες και πολλά στοιχεία δεν τα μαθαίνουμε, τα μαθαίνουμε ε, πλαγίως με στατιστικές από τα ασφαλιστικά ταμεία κτλ. Εδώ μπορεί να δώσει το παράδειγμα εκ την ιατρική στην ανθρώπινη ιατρική και να τη βάλει τα γυαλιά. Η χρήση αντιβιωτικών είναι τεράστιο πρόβλημα, αφορά όλου του τομεί τη κοινωνία και όλοι θα πρέπει να βοηθήσουν. Και στην κτηνιατρική και στην ανθρώπινη ιατρική. Από κοινού. Ευχαριστώ, κύριο Κέλλη. Ε, ε, Σας ευχαριστώ. ψήφισα για το κείμενο αυτό. Και με χαρά μου είδα ότι εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο. Θαυμάζω αυτόν τον ε, κλάδο. Νομίζω ότι η κοινωνία τους, δεν τους έχει εκτιμήσει όσο τους ε, αξίζει. Όπως είπε ο κύριος Γιάρ, ε, θεωρείται ότι τα πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε καλή φήμη όσον αφορά την λασιμότητα και ανιχνευσιμότητα για όλη τη διαδρομή του προϊόντος από το αγρόκτημα μέχρι το τραπέζι οπότε σήμερα ευτυχώς που πέρασε αυτό το κείμενο και έτσι θα εφαρμοστούν οι κανόνες το θέμα είναι ότι δεν τα πράγματα πάντα όπως τα θέλουμε άρα θα πρέπει με μεγάλη προσοχή να προστατεύσουμε την φήμη των ε, προϊόντων μας αλλά και την ε, φήμη του κλάδου αυτού που είναι παράδειγμα προς μίμηση. Ο Πρόεδρος. Και τώρα. Έχουμε το, το άλλο που αφορά μια που κάνουμε εδώ μερα κύριε Στάιλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ε, υπερψήφισα το ψήφισμα και ιδίω ε, ενδιαφέρομαι για αυτά που λέει για τις ψηφιακές δεξιότητες. Θα πρέπει τα κρατη μελινά συνειδητοποιήσουν τι δυνατότητες υπάρχουν. Θα πρέπει να συντονιστούν μεταξύ τους. Θα πρέπει να υπάρξει κατάλληλη παιδεία, κατάρτιση στο σχολείο, στις σχολές, στο πανεπιστήμιο. Παντού αυτό είναι κάτι που τώρα είναι πιο σημαντικό από ποτέ γιατί αν δεν υπάρχουν τέτοιες ψηφιακέ δεξιότητες δεν θα μπορέσει κανείς να εκμεταλλευτεί την ενιαία αγορά, να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης και να βοηθήσει την οικονομία. Χρειάζονται επομένω αυτές οι ψηφιακέ ε, δεξιότητε να διαπνέουν κάθε μας δραστηριότητα. Και ο Πρωθυπουργό αναφέρθηκε στην Κοινωνική Ευρώπη χθε και είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, τέτοια προσπάθεια τόσο ώστε κανείς Ευρωπαίος να μην μείνει πίσω, να μην μείνει εκτός αυτής της ψηφιακής επανάστασης. Και εγώ σας ευχαριστώ, λέω πρώτη, να στον κύριο Μαμίκης. Ευχαριστώ. 16-3 ε, δεδομένα θα έχουμε ε, ε, κάθε χρόνο, διότι η αύξηση των δεδομένων είναι 60% κάθε χρόνο. 40 bytes πάνω από 5.200 gigabyte ανακάτοικο αυτού του πλανήτη. Είναι τεράστιο το δυναμικό και θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Γι' αυτό και υποστηρίζουμε αυτή την έκθεση. Οι καταναλωτές, οι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, της παιδείας μπορούν να αξιοποιήσουν αυτό το δυναμικό. Χρειαζόμαστε πληροφορίες η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσουν τη χρήση, τη χρήση των μαζικών δεδομένων και όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό και ε, περιφερειακό και τοπικό. Ευχαριστώ. Κέλλη. Ε, ευχαριστώ. Άκουσα με ενδιαφέρον Είδα μάλλον, διαπίστωσα με ενδιαφέρον ότι υπήρχε μόνο μία εξαίρεση στον κατάλογο ψηφοφορίας και δεν ξέρατε ούτε κι εσείς ε, αν ε, ήταν οι βουλευτές υπέρ ή κατά. Πρόκειται για την τροπολογία 26 και νομίζω ότι δεν είναι σωστό αυτό. Δηλαδή τελικά χρειαζόμαστε ε, αποδείξεις και τεκμηρίωση για το πώς ψήφισαν οι άνθρωποι για όλες τις εκθέσεις, πώς ψήφισαν, πώς ήταν υπέρ, κατά, πώς απήχαν για όλες τις εκθέσεις. Είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση. Και νομίζω ότι είναι με καλή ευκαιρία για να προχωρήσουμε, να προοδεύσουμε σε αυτό τον τομέα. Πρόεδρος. Ξέρετε, οι πολιτικέ ομάδε ζητάνε την ε, ονομαστική ψηφοφορία. Εγώ απλώς εφαρμόζω τους ε, κανόνες. Και όχι, μα δεν ήμουν επικριτικός. Πιστεύω απλώς ότι θα πρέπει για τα πρακτικά ε, να υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες για όσους θέλουν να ξέρουν Ποιο ψήφισε τι. Ε, πρόεδρο, ναι, υπάρχουν κάποιε εκθέσει που θα άξιζε να έχουμε τέτοιε πληροφορίε. Λοιπόν, περνάμε τώρα στι προτάσει ψηφίσματο. Ερυθρέα. Πώ πιτσίλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υποστήριξα αυτό το ψήφισμα για την κατάσταση στην Ερυθρέα. Είναι τραγική η κατάσταση σε αυτή τη χώρα. Είναι από τις φτωχότερες χώρε αυτού του πλανήτη. δικτατορία. με ένα στρατό που έχει αμφίβολο ρόλο μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα προσπαθούν να ξεφύγουν ε, από τις εμπόλεμες ζώνες. Θα πρέπει να ζητήσουμε από την κυβέρνηση, από τον πρόεδρο να τηρήσουν ε, το διεθνές δίκαιο και νομίζω ότι αυτό μπορούμε έτσι να επηρεάσουμε την συμπεριφορά αυτού του δικτατορικού καθεστώτος. Ε, μπορούμε να αμφισβητήσουμε τη δράση τους και ελπίζω ότι θα ακολουθήσουν τις συστάσεις μας. Μαμίκινς, ευχαριστώ πρόεδρε. Η Ερυθρία σήμερα είναι σε ικτρή κατάσταση σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία της έκφρασης, ε, τους πόρους γενικά. Δεν υπάρχει ελεύθερο δικαστικό σύστημα και ανεξάρτητο. Και ο κάθε Ερυθρέος ηλικίας 18 με 50 ετών, με 50 ετών θα πρέπει να υπηρετήσει στο στρατό με ελεηνές συνθήκες. Γι' αυτό οι περισσότεροι ε, ε, φεύγουν από τη χώρα και γίνονται πρόσφυγες. Είναι βεβαίως αφρικανική χώρα ε, η Ερυθρέα γεωγραφικά, αλλά δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία δυνατότητα να επηρεάσει την κατάσταση στην Ερυθρέα. Δεν μπορεί δηλαδή να της πει να φέρεται καλύτερα. Και η κυβέρνηση σήμερα δεν δίνει δεκάρα για αυτά που λέμε εμείς εδώ. Ενώ ταυτόχρονα έχουν και πάρα πολύ κακές σχέσεις με τους γείτονές τους. Το ψήφισμα νομίζω θα βοηθήσει. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Κέλλη, υποστηρίζω απολύτως το ψήφισμα που έχει ε, υποβάλει δική μου ομάδα. Ε, σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση, στην Ερυθρέα καλούμε τις οι ευρωπαϊκές αρχές ε, καλούν ε, τη χώρα να αφήσουν ελεύθερους τους κρατουμένους, να χαλαρώσουν το καθεστώς ε, στρατιωτικής θητείας, να προχωρήσουν σε κοινωνικές παροχές, στέγαση κτλ. Ε, το δικαίωμα στην παιδεία επίσης να γίνεται σεβαστό ε, ε, πάρα πολλοί Ερυθρέοι εργάζονται να φύγουν από τη χώρα ακριβώ γιατί δεν γίνονται σεβαστά αυτά τα δικαιώματά του. Η ειρήνη και η ευημερία δεν νοούνται χωρί σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το κόμμα μου θα ήθελε να εκφράσει βαθιά ανησυχία για την έλλειψη ελευθερία τη έκφραση και τη συνεχιζόμενη ύπαρξη ε, πολιτικών κρατουμένων. Δεν γίνονται σεβαστέ οι αρχέ του κράτου δικαίου. Θα πρέπει να βυθούν να φυθεί ελεύθερος ο Ντέβι Τάζακ που είναι Σουηδο-Ερυθρέος και έχει ε, φυλακιστεί από το Σεπτέμβριο του 2001 χωρίς δίκη ουσιαστικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα θα περάσουμε στην επόμενη έκθεση που είναι έκθεση προόδου 2015 για τη Μακεδονία. Λέω πρόεδρος, ο λόγο και ο κύριος Πόσπιση. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα, ξέρετε, την έκθεση αυτή που παρουσιάζει την ε, παρούσα κατάσταση στη Μακεδονία, λέει ο μιλητής και αφορά την ε, διαδικασία ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι πεπισμένος ότι θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στη χώρα αυτή και στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων γενικότερα ε, μακροπρόθεσμα και για τη Μακεδονία συγκεκριμένα χαίρομαι πάρα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το προσφυγικό και την κρίση και πώς φυλάσσει και προστατεύει τα σύνορα. Ενώ η Ελλάδα έχει σταθεί ανίκανη να ε, ε, ελέγξει. Γι' αυτό θέλω να δω τη Μακεδονία ε, και να τη βλέπω ως σημαντικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώ η Ελλάδα μπλοκάρει την ένταξή της λόγω του ονόματος και νομίζω ότι αυτά τα μικρο θέματα δεν θα πρέπει να είναι καθοριστικά για το αν θα ενταχθεί μια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι, συγκεκριμένα η Μακεδονία. Ο Μαμίκινς. Ευχαριστώ Πρόεδρε η Βοσνία Ριζικοβίνη αλλά και η Τουρκία βρίσκονται στριμωγμένες όσον αφορά τις συνομιλίες ένταξης. Το ίδιο ισχύει και για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά με την Ελλάδα. Υπάρχουν εντάσεις και με την Βουλγαρία. Δεν είναι βέβαια αυτοί οι μόνοι λόγοι που δυσκολεύουν τις επαφές με την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς το παρόν δεν έχουν αρχίσει οι επαφές λόγω του Συμβουλίου. Πάντως το θέμα είναι ότι υπάρχει και πολιτική αστάθεια, υπάρχει διαφθορά. Δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου. Δυστυχώς δεν σημειώνεται πρόοδος στην υπόθεση. Ψήφισα το κείμενο αυτό και ελπίζω να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Ο επόμενος, ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ και πάλι. Ψήφισα και η πολιτική μου ομάδα υπέρ, αλλά όχι την τροπολογία 70 που αναφέρεται στο ΝΑΤΟ. Η Ιρλανδία είναι ουδέτερη χώρα, γι' αυτό και απέσχον. Πάντως με την ευκαιρία θα σα πω ότι συμφωνώ με τις άλλες ε, τροπολογίες. Νομίζω ότι η Μακεδονία θα σεβαστεί τις ευθύνες της και ότι θα υλοποιήσει όσα πρέπει με έναν τρόπο σοβαρό, συνεχή, συνεπή και θα μπορέσει να ανοίξει τα κεφάλαια της διαπραγμάτευσης που κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και συμφωνώ με την Επιτροπή Άφετο ότι θα πρέπει να υπάρχει επικοδομητικός διάλογος γιατί έρχονται εκλογές στις 5 ε, Ιουνίου του 16 και σας ευχαριστώ. Μακοβέη. Μάλιστα, είναι αλήθεια ότι η Μακεδονία αντιμετωπίζει από το 2001 την πιο σοβαρή κρίση της ιστορίας της. Επομένως οι προσπάθειες της χώρας κατατείνουν στην έξοδο από αυτή την κρίση. Χρειάζεται να βρει η κοινωνία τη σταθερότητα και να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην το ξεχνούμε αυτό. Ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εντολή των διαπραγματεύσεων από το Συμβούλιο. Όμω το Συμβούλιο είπε όχι γιατί έχει αντίρρηση η Ελλάδα. Νομίζω ότι θα πρέπει και η Ελλάδα να αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλει η χώρα. Επίσης καταβάλει προσπάθεια και για το προσφυγικό. Είναι σημαντικά τα μέτρα που έλαβαν οι αρχές της χώρας. Χρειάζεται την ε, βοήθειά μας. Και έτσι θα τηρήσουν τις υποσχέσεις τους και αν δεν κάνουμε θα το πιατάζουμε θα χάσουμε αξιοπιστία. Και τώρα έχουμε την έκθεση για το Μαυροβούνιο. Ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας. Το Μαυροβούνιο άρχισε διαπραγματεύσεις για την ένταξη του στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από μία τετραετία και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Η Ευρώπη όμως θα πρέπει να επιταχύνει Πέρυσι ήταν θετικά τα αποτελέσματα και σε άλλους τομείς στην εφαρμογή του κράτους δικαίου μπορεί οι βελτιώσεις να μην είναι τόσο θεαματικές ούτε τόσο ταχείες όσο εμείς θα επιθυμούσαμε ή θα αναμέναμε αλλά ε, είναι θετικές εξελίξεις εν γέννη. Επίσης το εκπαιδευτικό σύστημα έχει μεταρρυθμιστεί και το εκτιμώ πάρα πολύ όπως και την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κέλλη. Πρόεδρε, και πάλι ε, πρέπει να σας πω ότι μαζί με την ομάδα μου υπερψήφισα την έκθεση για το Μαυροβούνιο και δεν δυσκολεύτηκα ε, γιατί είναι πολύ θετικές οι εξελίξεις. Το Μαυροβούνιο ε, έχει τους υψηλότερους βαθμούς ανάπτυξης από τις γύρω χώρες και ελπίζουμε σύντομα να το καλωσορίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέλος. Είναι πολλές οι χώρες που θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλες όπως η Βρετανία προσπαθούν να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ταυτόχρονα ας αναγνωρίσουμε ότι έχει σημειώσει με τα πρόοδο το Μαυροβούνιο και όσον αφορά τα δικαιώματα των ε, γυναικών. Άρα ε, οπωσδήποτε πρέπει να αναγνωρίσουμε το ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ακόμα μεταχείριση. Θα πρέπει επίση να καταπολεμηθεί η φτώχεια στην ε, χώρα και έτσι να γίνει ε, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρία Μακοβέη, το Μαυροβούνιο έχει ανοίξει 22 διαπραγματευτικά κεφάλαια. Μερικά ημέρα έχουν κλείσει σημαντικό βήμα ένταξη. Άρα να τονίσουμε το ότι έχει καταβληθεί προσπάθεια καταπολέμηση τη τρομοκρατία από την κυβέρνηση. Επίση ε, έχουν ε, καταπολεμήσει του τζιχαντιστέ. Και βέβαια το πρόβλημα τη χώρα είναι η διαφθορά θα πρέπει να υπάρχει κώδικα διοντολογία για του ε, δικαστέ. Αυτό θα αλλάξει τα πράγματα γιατί δεν είναι αναγκαστή κανόνες δικαίου αυτά. Δεν, δεν, δεν προβλέπονται κάποιες κυρώσεις. Ε, θα πρέπει να υπάρξει καταδίκη ε, της τη διαφθορά, θα πρέπει να γίνονται κατασχέσει, θα πρέπει να, γίνουν, να ανοίξουν οι φάκελοι και θα πρέπει επομένω να θεσπίσουν κάποια νομοθεσία πιο βαριά και να προβλέπει και οι κυρώσεις. Μόνο επομένως ε, έτσι και με βαριές ποινές θα καταπολεμηθεί η διαφθορά. Το ίδιο ισχύει και για το οργανωμένο έγκλημα, αλλά και για το ξέβλημα χρήματος. η ε, η λύση προβλήματος στο Μαυροβούνιο και θα πρέπει να δείξουν ε, αποφασιστικότητα, ώστε να μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημα. Και τώρα ο κύριος Μάμπικινς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το 2012 από ό,τι ξέρουμε, σαν αντιδράσει την κρίση, και αρχίσαμε να εφαρμόζουμε τη νέα πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρχισε η ρύθμιση σε υπερεθνικό επίπεδο για τον τραπεζικό τομέα και εγώ καλωσορίζω όλα τα βήματα που έχουν γίνει. Θα ήθελα να επιταχυνθούν οι διαρθρωτικές αλλαγές στο τραπεζικό τομέα ώστε να γίνει αθεκτικότερος για μελλοντικές κρίσεις. Κυρίως μιλώ για τις big banks, τις μεγάλες συστημικές τραπεζές. Νομίζω ότι όλοι θα κερδίσουμε από αυτή τη νέα ρύθμιση, διότι για τους καταθέτες θα έχουν εγγυημένες καταθέσεις τους, παραδείγματο χάρη, θα προβλέπεται αποζημίωση ανεξαρτήτως από την τοποθεσία της τράπεζας. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Στάκουλα. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ καταψήφισα αυτή την έκθεση για την Τραπεζική Ένωση. Εγώ θεωρώ πως ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχουν ε, πλεονεκτική θέση σε σχέση με τους φορολογουμένους και τους καταθέτες ε, που ε, αναγκάζονται να πληρώσουν τα σπασμένα σε περίπτωση κρίση. Έχουμε πολλαπλά παραδείγματα από τα προηγούμενα χρόνια και έχουμε φτιάξει μια κοινή ένωση χρέους, όχι τραπεζική ένωση. Εγώ όμως είμαι φιλοευρωπαίος και θέλω να αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή συνεργασία. Όμως ε, νομίζω ότι με τέτοιου είδους δομές θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα ευέλικτο σύστημα, ένα υγιές τραπεζικό σύστημα ε, και να από το αποσυνδέσουμε από τις υπόλοιπες δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε και πάλι και συγχαρητήρια. Είστε αποτελεσματικότερο στην Προεδρία, συγγνώμη, στην Προεδρία. Και ε, καταφέρνετε να διατηρήσετε το χιούμορ σας ενώ είναι δύσκολο σε αυτό τον τομέα με αυτά που συνέβησαν σε περίπτωση οικονομικής ύφεσης και σε χώρες όπως και η δικιά μου. Και ε, Χαίρομαι ιδιαίτερω από την εποπτεία τραπεζών να αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουμε τεστ κοπόσεω και ούτω καθεστώ και κανόνε που ισχύουν σε όλη την επικράτεια τη Ένωση. Διότι σε μια μικρή χώρα όπω η Ιρλανδία είναι πολύ εύκολο να έχουμε καταχρηστικέ πρακτικέ και να υπερασπίζονται τα συμφέροντα μόνο των πλουσίων. Ε, να η ευκαιρία για μια ουσιαστική ένωση με ε, κατάλληλη τραπεζική διαχείριση και δεν θα χρειάζεται να πληρώνουν το μάρμαρο οι ε, καταθέτες και οι και ελπίζω το too big to fail να εκλείψει ως αρχή. Ε, ελπίζω ότι βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διαχειριζόμαστε τις τράπεζες και πρέπει οι ίδιοι οι κανόνες να ισχύουν για τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε κύριε Κέλλη. Ευχαριστώ διπλά κύριε Κέλλη και για τις φιλοφρονήσεις. Συνάδελφοι, η χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε από το 2007 και έχει κάνει άνω κάτω όλο το δυτικό κόσμο δείχνει ότι οι πολιτικοί θέλουν ε, να ε, βγάλουν το ρίσκο ε, από τη Μέση Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει την ευκαιρία και όπως κάνει πάντα την έχει πιάσει η μεγαλομανία της θέλει να πέρασει στην τρίτη φάση της εγγύησης των καταθέσεων και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αυξηθεί ο κίνδυνος να είναι η ένωση, μια ένωση μεταφοράς πόρων από το βορρά προς τον νότο και είμαστε σε μια κλιμάκωση και χωρίς τέλος. Γι' αυτό σήμερα εγώ καταψήφισα την έκθεση Γκουαλτιέρη. Ευχαριστώ κυρία Γκραπίνη. Ε, Κύριε Πρόεδρε, εγώ υπερψήφισα την έκθεση γιατί πιστεύω ότι χρειαζόμαστε την Τραπεζική Ένωση ε, και αυτό θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην χρηματοδότηση ε, των επενδύσεων για τις μικρομεσαίες. Εάν μειώσουμε ε, το κίνδυνο των τραπεζών τότε θα ε, μειωθεί και το κόστος χορηγήσεων. Χρειάζεται ενιαίος εποπτικός μηχανισμός με ποιοτική εποπτεία και όχι υπερβολική ε, προληπτική διαχείριση ε, και να περάσουμε, να μετακυλίουμε το κόστος όλο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι χορηγήσεις και τα δάνεια στις μικρομεσαίες είναι ζωτικής σημασίας και δεν θα πρέπει να μπλοκάρουμε τη νέα τεχνολογία, την έρευνα και την καινοτομία. Χαίρομαι που αναλαμβάνει ευθύνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την έκθεση γιατί πρέπει να εξασφαλίζει το θεμητό ανταγωνισμό. Ευχαριστώ. Ε, διακοπή της συνεδρίασης μέχρι τις 3 λέει ο Πρόεδρος.